για την ασφάλεια στην Ευρώπη. Ευχαριστώ, Επιτροπέ Oettinger. Και τέλος, ε, κατατέθηκε ένα ψήφισμα από την Επιτροπή ε, Βιομηχανίας. Αύριο στις 12 θα ψηφίσουμε. Ολοκληρώνεται λοιπόν η συζήτηση και έχουμε μια κοινή συζήτηση για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και έχουμε καταρχάς την έκθεση του κυρίου Αρσένη, Λογιστική Κανόνα και σχέδια Δράση για τι εκπομπέ και τι απορροφής αερίων θερμοκηπίου. Και έχουμε και την έκθεση ICOUT, μηχανισμό παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων σχετικά με τι εκπομπέ αερίων θερμοκηπίου και υποβολή άλλων πληροφοριών που αφορούν την κλιματική αλλαγή. Καταρχά θα ακούσουμε του δύο εισηγητέ. Καταρχά, τέσσερα λεπτά ο κύριο Αρσένη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Συντάμε για δύο συγκεκριμένε εκθέσεις, την έκθεση για το ΛΟΥΣΙΕΦ και το MRV και το MRR, αλλά σε κάθε περίπτωση το θέμα που συζητάμε εδώ πέρα είναι η κλιματική αλλαγή. Κάθε χρόνο συναντιόμαστε στις κλιματικές διαπραγματεύσεις. Κάθε χρόνο σημειώνεται πρόοδος. Όμως κάθε χρόνο, χρονιά μετά από τη χρονιά, συνεχίζει αυτή η πρόοδος να μην είναι ικανοποιητική, να μην είναι αρκετή προκειμένου να έχουμε σημαντικές πιθανότητες να πετύχουμε την, κλιματική, Παγκόσμια Κλιματική Συμφωνία μέχρι το 2015. Τι κάνουμε λάθος, τι είναι αυτό που πρέπει να αλλάξει. Μέσα από τις δύο αυτές εκθέσεις η άποψη του Κοινοβουλίου είναι σαφής. Πρέπει να αλλάξουν οι ρυθμοί μας και η αποφασιστικότητά μας, η σοβαρότητά μας και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Χρειάζεται όταν γυρνάμε ε, από τις διεθνείς διαπραγματεύσεις όχι απλά να μεταφέρουμε τις διεθνείς αποφάσεις στην ευρωπαϊκή νομοθεσία αλλά να τις πηγαίνουμε πολλά ε, βήματα παραπέρα να τις ολοκληρώνουμε. Αυτό και κάναμε με το LULUCF. Ακριβώς μετά την, τον Τέρμαν ήρθε η πρόταση της Επιτροπής ε, για την εσωμάτωση της απόφασης του Ντέρμπαν για τις υπολογισμό των εκπομπών, καταγραφή των εκπομπών από τη χρήση και αλλαγή χρήση γης. Αντί όμως αντί να παραμείνουμε στο ελάχιστο που είχε αποφασιστεί στο Ντέρμπαν, στις κλιματικές διαπραγματεύσεις, την υποχρέωση για καταγραφή των εκπομπών που προέρχονται από τα δάση, είτε είναι η αναδάσωση, είτε είναι η δάσωση, είτε είναι η διαχείριση των δασών και άλλα, προχωρήσαμε παραπέρα. Κάναμε υποχρεωτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη και την καταγραφή των εκπομπών που αφορούν τις γεωργικές δραστηριότητες. Και όχι μόνο αυτό. Μέσα στην ομοθεσία έχουμε την υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να πρωτοστατήσει στις κλιματικές διαπραγματεύσεις προκειμένου σε διεθνέ επίπεδο να γίνει υποχρεωτική και η καταγραφή των ε, εκπομπών και ο υπολογισμό των εκπομπών που προέρχονται από του υγροτόπου. Και νομίζω ότι με τον τρόπο αυτό, αν συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, αν πραγματικά σοβαρέψουμε ε, τις πολιτικές μας, αν κάνουμε τις πολιτικές μας πιο υπεύθυνε, θα μπορέσουμε να φτάσουμε το 2015 σε μια παγκόσμια κλιματική συμφωνία που τόσο χρειαζόμαστε. Όμως δεν δεν επιτυχάνονται ε, αυτές οι πρόοδοι αυτόματα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πέρα από όλους τους συναδέλφους, ε, τις σκιώδεις εισηγητές αυτήν την έκθεση που στηρίξαν την εισαγωγή των γεωργικών εκπομπών στο να είναι υποχρεωτικά ε, να καταγράφεται υποχρεωτικά κάθε χρόνο, όπως θα συμβαίνει από εδώ και μπρος. Θέλω να ευχαριστήσω τον συνεργάτη μου που ασχολήθηκε με αυτό το θέμα, Λία Πρέβεζα, την ε, Ulrike Σόνερ ε, από την, Γραμματεία των Σοσιαλιστών, την Σύμβουλο Σοσιαλιστών σε αυτά τα θέματα, την Ιζαμπέλ Φίντλεϊ από την Γραμματεία της, ε, της Επιτροπής Περιβάλλοντος, την Κυπριακή Προεδρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλοι μαζί καταφέραμε με διαδικασίες εξπρές να ολοκληρώσουμε την, σε πρώτη ανάγνωση αυτή τη διαπραγμάτευση και ήδη από το 2013 να αρχίσει η καταγραφή των ε, αγροτικών εκπομπών από τα κράτη μέλη. πρέπει να καταφέρουμε μέχρι το 2015 να έχουμε την κλιματική, παγκόσμια κλιματική συμφωνία και θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ συνάδελφε Αρσένη. Για τέσσερα λεπτά ο κύριος Άικαουτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντα ε, τους κοιόδη εισηγητές στην Επιτροπή και την Κυπριακή Προεδρία για τη συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Αυτό δεν θα είχε επιτευχθεί αν δεν είχαν κάνει όλοι ό,τι καλύτερα μπορούσαν. Η, εισήγηση, η έκθεση στην οποία ήμουν εισηγητής ήταν πάρα πολύ σημαντική σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις που έχουν τα κράτη-μέλη για τα εκπομπές αερίων θερμοκηπίου προκειμένου όλοι να ακολουθούν τους ίδιους κανόνες με την ίδια διαφάνεια σε ό,τι αφορά τα αέρια αυτά. Αυτό που είναι σημαντικό και ιδιαίτερα σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να μας υποβάλλουν στοιχεία για την μετάβαση της οικονομίας σε μια οικονομία η οποία θα μειώσει κατά 80-90% των αερίων θερμοκηπίου. Αυτό μπορεί να ακούγεται ως μακροπρόθεσμο στόχος, αλλά αυτές οι αλλαγές θα πρέπει να γίνουν σύντομα και αυτή η έκθεση καταδεικνύει τα επόμενα βήματα. Ένα άλλο σημαντικό θέμα ήταν η ναυτιλία, οι θαλάσσιες μεταφορές, γιατί αυτό φαίνεται ότι δεν το αποδέχονται τα κράτη-μέλη, δεν το συζητάνε καν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ε, θέλει να υποβάλει σχετικές προτάσεις και ανυπομονώ να τις ακούσω αυτές τις προτάσεις προκειμένου να έχουμε μια σαφή βάση. Το πιο σημαντικό σημείο και το σημείο το οποίο εξετάσαμε πιο πολύ στις ε, διαπραγματεύσεις είναι οι υποχρεώσεις ε, αναφοράς υποβολής εκθέσεων σε ό,τι αφορά τα χρηματοοικονομικά στοιχεία και θα ήθελα να τονίσω ότι οι δύο κράτη-μέλη τα οποία προβάλλουν το πράσινο χαρακτήριο, αλλά δυσκόλυψαν πάρα πολύ τι διαπραγματεύσει. Η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ήταν πάρα πολύ περίεργο αυτό, ακόμα και σε ό,τι αφορά τι υποχρεώσει υποβολή εκθέσεων για το πόσα χρήματα δίνουμε στην υποστήριξη του κλίματο, Ακόμα και αυτή η υποχρέωση ήταν τεράστιο πρόβλημα για το Ηνωμένο Βασίλειο και για την Γερμανία. Άρα, σε κάθε ευκαιρία παρουσιάζονται ως οι πιο πράσινες οικονομίες, αλλά τελικά όταν τους ζητάμε να μας πούν πόσα χρήματα δίνουν στις αναπτυσσόμενες χώρες μας ε, άρουν εμπόδια μόνο και μόνο επειδή δεν θέλουν να ε, δώσουν τέτοια στοιχεία. Να σας ε, πω ότι η έκθεση αυτή δεν έχει να κάνει με τις αρμοδιότητες των κρατών μελών. Αυτό που ζητάμε είναι να υποβάλλεται έκθεση για το πόσα χρήματα δαπανούνται κάθε χρόνο στις αναπτυσσόμενες χώρες. Και ξέρουμε πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την υποστήριξη του κλίματος. Κάθε χρόνο είναι τεράστια η μάχη που δίνουμε και κάθε φορά, κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να ξεκαθαρίσει πόσα χρήματα θα πανά προς την κατεύθυνση αυτή, γιατί δεν το λένε τα κρατή-μέλη, όπως και την προηγούμενη φορά στην Τόχα, η Δανία έδωσε κάποια στοιχεία, μάλλον ε, η Δανία, η Σουηδία, η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, δαπανούν χρήματα, αλλά δεν μπορούμε να παρουσιάσουμε ένα άθροισμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά τα χρήματα που δίνουμε στις αναπτυσσόμενες χώρες. Και αυτό είναι κάθε χρόνο ένα πρόβλημα στις διεθνείς διαπραγματεύσεις. Και χάρη στην έκθεση αυτή θα πάρει τέλος αυτή η κατάσταση. Αλλά πραγματικά τεράστια αντίσταση αντιμετωπίσαμε από το Ηνωμένο Βασίλειο και από τη Γερμανία. Είναι σημαντικό λοιπόν κράτη-μέλη αυτά που κάνετε για το, το, κλίμα είναι όλα σημαντικά, αλλά ας φροντίσουμε να έχουμε και μια δύναμη σε Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί το θέμα εδώ πέρα στην έκθεση αυτή ήταν η υποβολή έκθεση. Αν και αυτό μας δυσκολεύει, τι να πω. Είναι μακρύς ο δρόμος για μια πραγματικά πράσινη οικονομία. Λοιπόν, έχουμε τις υποχρεώσεις πλέον για την υποβολή έκθεση και τώρα πραγματικά θέλουμε δράση. Ευχαριστώ, συνάδελφα. Και τώρα η Επιτροπός κάρτα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. My sincere appreciation for the two rapporteurs, Kriton Asinis and Bas Aykut. Και ευχαριστήσουμε τους εισηγητές, να ευχαριστήσουμε τους εισηγητές και την γραμματεία για αυτές τις δύο νομοθετικές προτάσεις και ε, με αυτόν τον τρόπο είχαμε μια συνεργασία πάρα πολύ παραγωγική ε, μεταξύ των θεσμικών οργάνων και επίσης ε, και η Κυπριακή Προεδρία βοήθησε πάρα πολύ και έτσι μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε με τη διαδικασία συμφωνώντας στην πρώτη ανάγνωση και για τα δύο κείμενα. Τώρα, μπορέσαμε τελικά να ε, κάνουμε ένα βήμα προς τα εμπρός, μπορέσαμε να καλύψουμε το όσα έχουμε ε, υποσχεθεί όσον αφορά την ε, πολιτική για το κλίμα και έτσι επομένως μπορούμε να πούμε να δείτε ότι κατά αυτόν τον τρόπο θα θέλουμε υπόψη τις τόσο που στον Τέρμαν και επίσης ε, έτσι ε, σύμφωνα με τη UNSC καλύπτουμε το ΝΑΟ και προς το 2020 ε, τις σχετικές, το σχετικό πρόγραμμα και επίσης καλύψαμε αυτόν τον τομέα στους εθνικούς λογαριασμούς των κρατών μελών και τώρα μπορούμε να γεφυρώσουμε αυτό το χάσμα οπότε και στο μέλλον μπορούμε όλους τους τομές να τους καλύψουμε όσον αφορά την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και κατά αυτόν τον τρόπο έχουμε κάποιες, κάποιες διασφαλίσεις για τη γη και σε σχέση με τόσο αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πάρα πολύ βασικές πτυχές της πρότασής μας βέβαια ήταν ο συνδυασμός οπότε έτσι θα έχουμε υποχρεωτική λογοδεσία από το 2020 και μετά όμως έχουμε και κάποια βαθμία προσέγγιση για αυτές τις δραστηριότητε κατά την περίοδο μέχρι το 2020. Όλα αυτά θα πρέπει να θεωρηθούν ότι είναι ένα πρώτο βήμα και έτσι μπορούμε τώρα να συλλέξουμε κάποια δεδομένα στις γεωργικές υγείες και τώρα μπορούμε επίσης να δούμε πώς τα κρατημέλη μπορούν να ενθαρρύνουν τις άριστες πρακτικές, να συλλέξουμε πληροφορίε και έτσι να μπορούμε να έχουμε καλύτερη ρύθμιση στον τομέα στο μέλλον. Με αυτή την πρόταση επίση μπορούμε να δούμε το ότι θα έχουμε μια οικονομία βιώσιμη. Και μπορούμε τώρα να προωθήσουμε κάποια συστήματα και μεθοδολογίες για να προστατεύσουμε την ύπεθρα και το έδαφος. Χρήση βιομάζας και άλλων ανανεώσουμε πηγών ενεργείας θα καλυφθούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης εάν γίνει γρήγορη εφαρμογή της απόφαση, τότε θα μπορέσουμε να μάθουμε καλύτερα τα προβλήματα και ταυτόχρονα να συζητηθεί το τι και πότε επιβάλλεται να γίνει. Το πρώτο άρθρο της Λουλούσεφ ορίζει ότι αυτό είναι μόνο ένα πρώτο βήμα. Το επόμενο βήμα αφορά το πώς και πότε αυτές οι εκπομπές μπορούν να περιληφθούν στη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση των εκπομπών. Είναι ένα ορόσημο, έρεται ένα κενό στην πολιτική μας και διευκολύνει πάρα πολύ τη συζήτηση. Σε σχέση με το τι ρόλο θα πρέπει να παίξει ο, τομ, ο τομέας αυτός στην κλιματική πολιτική. Για το MMR τώρα δύο λόγια. εδώ έχουμε την πρόταση της Κομισιόν, τόσο ώστε να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερο μηχανισμό υποβολής αναφορών. Επίσης έτσι έχουμε το Δημοτικό Παγιο του 2009, το οποίο ακολουθούμε και η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κρατημέλη συμμορφώνονται με τόσο που αποφασίστηκαν στο Κιώτο και τέλος μπορούμε να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε παρακολούθηση και υποβολή αναφορών και εκθέσεων για τις εκπομπές. Το κείμενο αυτό, όπως συμφωνήθηκε, θα καλύψει τους στόχους μας. Ξέρουμε ότι δεν τα λύσαμε όλα, δεν τα καλύψαμε όλα. Αυτό έχει να κάνει και με κάποια στρατηγική χαμηλών εκπομπών, χρηματοδότησης, συγνότητα έκθεσης και το τι θα γίνει με τις εφαρμοστικές πράξεις και ως τμήμα αυτής της συμφωνίας δεχθήκαμε προβλήματα σε δύο ανακοινώσει οι οποίες πρόκειται να σας διαβαστούν ούτως ώστε να τις περιλάβετε στα πρακτικά σας. Παρ' όλα αυτά, εμείς χαιρετίζουμε αυτό το συμβαστικό κείμενο. Έτσι μας δίνει τα μέσα που χρειαζόμαστε για να μπορέσουμε να είμαστε πρωτοπόρες στις παγκόσμιες προσπάθειες να παραμείνει η δημοκρασία κατά από τις δύο δύο βαθμούς, να ελαχιστοποιήσουμε τις αλλαγές του κλίματος και να είμαστε συμμορφωμένοι με τα όσα έχουμε υποσχεθεί διεθνώ και τα μέσα επόμενα χρόνια θα συνεργαστούμε το κράτος μέλος, με τα κράτη-μέλη, θα ενημερώνουμε το Κοινοβούλιο και θα παρακολουθούμε την εφαρμογή της ε, συμφωνίας MMR και θεωρούμε ότι τα έχουμε πολλέ εναλλακτικές για να ε, προχωρήσουμε καθώς και τη διαξία της συναπόφασης και κατακλείδη να σας πω ότι η αυριανή ψηφοφορία θα αποτελέσει μια επιτυχία και για τις δύο αυτές συμφωνίες και θα είναι πολύ σημαντικό βήμα αυτό που κάναμε εδώ. Κυρία Χίντεγκαρ, ε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχει σημειωθεί η υπέρβαση του χρονοδιαγράμματος ε, συνεδριάσεων και αυτό απευθύνω θερμή παράκληση το χρόνο ομιλίας. Ε, το λόγο έχει η συνάδελφος κυρία Βέστλουντ, εξ ονόμα της Επιτροπής Ανάπτυξης, για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Είναι σημαντικό να υπάρχουν ρυθμίσεις και κανόνες για τα στατιστικά στοιχεία και για την υποβολή εκθέσεων και να τηρούνται οι κανόνες αυτοί και σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις ε, για το κλίμα σε όλα τα πολιτικά επίπεδα. Γι' αυτό όντω είναι σωστό να γνωρίζουμε πόσα κράτη-μέλη ξοδεύουν τι ακριβώς για αναπτυξιακή βοήθεια. Όπως είπε και ο κύριος Άικχαουτ, ε, θα ζητήσουμε πιο πολλά συγκεκριμένα στοιχεία στις μελλοντικές συζητήσεις και θεωρώ ότι είναι κρίμα το γεγονός ότι ασκούμε τόσο πολύ κριτική στο σημείο αυτό. Τα χρήματα αυτά ε, ουσιαστικά φεύγουν από την ανθρωπιστική βοήθεια για να δαπανηθούν σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Ελπίζω να σημειωθεί πρόοδος στο σημείο αυτό σε ό,τι αφορά την ε, επιπλέον χρηματοδότηση ε, για θέματα κλίματο. Να μην αφαιρούνται τα χρήματα αυτά από την ανθρωπιστική βοήθεια. Ευχαριστώ. Δεν βλέπω στην αίθουσα του συνάδελφο κ. Χατζηγεωργίου. Έτσι ανοίγει ο κύκλο των ομιλητών εξ ονόματο των πολιτικών ομάδων. Το λόγο έχει εξ ονόματο τη ομάδα του ΕΛΚ η συνάδελφο κυρία Μορκινάιτε Μικουλιανένε. Για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χωρίς καμία αμφιβολία η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, βρίσκεται σε ηγετική θέση για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είμαστε αρκετά φιλόδοξοι ή κατά πόσο είμαστε μόνοι. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση των κλιματικών αλλαγών και το πρωτόκολλο του Κιώτο μας επιβάλλουν να αναλάβουμε αποφάσεις στον τομέα Λουλουσέφ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προβάλει ένα φιλόδοξο σχέδιο λαμβάνοντας ε, υπόψη και κανόνες λογοδοσίας. Θα πρέπει να επιβάλλουμε μέτρα κάποια χρονική στιγμή και γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την ε, αναλογικότητα, την αρχή της αναλογικότητας. Όταν μιλήσαμε για δοκιμές αντοχής, είπα ότι ο τομέας του Λουλουσεφ δεν θα πρέπει να αποτελεί επιπρόσθετο φόρτο για τα κρατη ή τους αγρότες και δεν θα πρέπει να επιφέρει και επιπρόσθετες υποχρεώσεις έτσι ώστε να μην ε, υπάρχει λογοδοσία. Ο τριμερής διάλογος ε, κατασύγασε τις βασικότερες ανησυχίες μας και μιλάμε για μέτρα που λαμβάνονται και μέσα στα πλαίσια της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών. Αλλά ως προς τη δασοκομεία δεν έχουν ε, ληφθεί ακόμα οριστικές αποφάσεις. Ελπίζω να μην αποτελέσει αυτό πρόσκομα για τη μελλοντική μας πορεία. Εξ ονόματος της ομάδος S&D το λόγο έχει η συνάδελφος κυρία Ουλφσκοκ για δύο λεπτά. Ε, Ευχαριστώ πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά την πολιτική για το κλίμα, βλάπτεται σημαντικά από, την... από τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των κρατών μελών Και αυτό τελικά μας οδηγεί σε μία απραξία, γιατί δεν μπορούμε να λάβουμε αποφάσεις. Αυτές οι ασυμφωνίες μεταξύ κρατών μελών είναι πολύ δύσκολες. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να γνωρίζουμε ακριβώς ποια αποτελέσματα έχουμε πετύχει. Αυτή η υποχρέωση για την υποβολή εκθέσεων προκύπτει από τη δυσκολία που έχουμε για τη συγκρισιμότητα των στοιχείων. Και ο εισηγητής υποστηρίζει λοιπόν την κατεύθυνση αυτή. Η πρόταση επιτρέπει εκθέσεις από πλευράς των κρατών μελών, οι οποίες αφενός θα έχουν ε, να κάνουν με την ε, προστασία του κλίματος και την χρήση των ανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ε, θέλουμε η κλιματική πολιτική να εφαρμοστεί και στην πράξη. Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε τις προσπάθειες αυτές. Ευχαριστώ πολύ. Ε, ο, ο συνάδελφος ε, κύριος ε, Ζιόμπρο θέλει να κάνει χρήση της μπλε κάρτας. Αποδέχεις το αίτημά του. Παρακαλώ, κύριε Ζιόμπρο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να υποβάλω μία ερώτηση Όσον αφορά τις κλιματικές αλλαγές, θα ήθελα να σας ρωτήσω ως εκπρόσωπο των σοσιαλιστών κατά πόσο υπάρχει σχέση αιτιόδου συνάφειας στη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μία ε, οικονομία με χαμηλή κατανάλωση άνθρακα. Υπάρχουν μεγάλες επιχειρήσεις που μετακινούνται μετεγκαθίστανται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκεί όπου δεν υπάρχουν περιορισμοί ε, εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, όπως στην Ασία. Και έτσι η Ευρώπη χάνει. Εσείς είστε σοσιαλιστής, γι' αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς το αποτιμάτε. Det här är en del av eh, klimatdiskussionen eh, i allra högsta grad. Eh, Βεβαίως, οι κλιματικές αλλαγές διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο και οπωσδήποτε θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για την εξέβρεση παγκόσμιας συμφωνίας για να μην μετεγκαθίστανται επιχειρήσεις αλλού με αλγινές συνθήκες εργασίας και μεγαλύτερες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Αυτό το βλέπω από πλευράς Επιτροπής Περιβάλλοντος αλλά και Επιτροπής Βιομηχανίας. Υπάρχει και το στοιχείο του ανταγωνισμού. Γι' αυτό θα πρέπει να δράσουμε ευφυώς. Σώματος της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη, το λόγο έχει ο συνάδελφος κ. Θεόδωρος Χιλακάκης για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, οι εκθέσεις αυτές έχουν τεχνικό χαρακτήρα και στα βασικά στοιχεία του πετύχαμε πιστεύω έναν καλό συμβιβασμό. αναδεικνύουν όμως και πολύ σοβαρά πολιτικά θέματα καθώς οθούν προς μεγαλύτερη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα σε ό,τι αφορά την κλιματική μας πολιτική. Και χρειαζόμαστε πράγματι στην κλιματική μας πολιτική και μεγαλύτερη διαφάνεια και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Στο πλαίσιο του ETS, του εμπορίου ρήπων για παράδειγμα, άνθησαν δυστυχώς σοβαρά σκάνδαλα το πιο μεγάλο σε μέγεθος ήταν το σκάνδαλο των cdm για τον τερματισμό του οποίου έδωσε μάχη η επίτροπος η ίδια αλλά έδωσε μάχη και το κοινοβούλιο και βοήθησα μπορώ να σας πω και ο ίδιος. και η αντίδρασή μας η κοινή αυτή οδήγησε στην εξοικονόμηση εκατοντάδων εκατομμυρίων ή και δισεκατομμυρίων ευρώ για τον ευρωπαίο καταναλωτή ηλεκτρικού ρεύματος αφού προηγουμένως είχαν πληρωθεί αντίστοιχα ποσά σε εργοστάσια εκτός ευρώπης και ενδιάμεσους που κερδοσκόπησαν αξιοποιώντας την πολυπλοκότητα και διαφάνεια του συστήματος πουλώντας μας δικαιώματα μέχρι και 70 φορές ακριβότερα από ό,τι είχαν κοστίσει. Αντίστοιχα, χρειαζόμαστε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα έτσι ώστε να μην επαναληφθεί και το φαινόμενο των φωτοβολταϊκών πάνελ που τα αγοράσαμε πανάκριβα για να δημιουργήσουμε μια ισχυρή ευρωπαϊκή πρωτοπορία και είδαμε στο τέλος την κίνα να μας παίρνει την αγορά επιδοτώντας απευθείας τους δικούς της παραγωγούς για να αποσπάσει τις επιδοτήσεις που εμείς δίναμε όλα αυτά τα χρόνια. Τα λάθη αυτά ελπίζω να αποφευθούν στο πλαίσιο του LULUCF, όπου από την αρχή εξασφαλίζονται ικανοποιητικοί πιστεύω κανόνες λογιστικής απεικόνησης. Θα το δούμε όμως στην πράξη και θα είμαστε πάντα σε εγρήγορση υπερασπιζόμενοι τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα στην κλιματική μας πολιτική. Γιατί το θέμα είναι πολύ μεγάλο και πολύ κρίσιμο για να το αφήνουμε έρμεο μόνο στα ωραία λόγια και στις καλές προθέσεις. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ τον συνάδελφο κ. Χιλακάκη. Εξ ονόματος ομάδας των Προσύνων, καλώ στο βήμα τη συνάδελφο κυρία Χάση. Για ένα λεπτό. Hyvät kollegat, kiitos raportööreille erittäin hyvästä ja omistautuneesta työstä. Ευχαριστούμε τους συγητές για την εξαίρετη εκθεσή τους. Ξέρετε, σε όλο τον χρόνο τα δάση και η γεωργία ευθύνονται για το εν πέμπτον του συνολικού εκπομπών. Όπως και οι μεταφορές πάρα πολλοί θεωρούν ότι η γεωργία αλλά και τα δάση μειώνουν τις εκπομπές όμως. Έχουμε πάρα πολλές πρακτικές που είναι φιλοπεριβαλλοντικές όμως και πάρα πολλές παραδοσιακές πολιτικές που πρέπει να τεθούν ένα αμφιβόλο. Αυτό ισχύει και τη δική μου χώρα. Εάν δεν χρησιμοποιήσουμε τις καλύτερες από τις πρακτικές, εάν δεν κάνουμε τις σωστές αναφορές και εκθέσεις, τότε θα πάνε χειρότερα. Ας πούμε, δεν θα πρέπει να έχουμε τα, το, το μέρος που είχε τύρφη να το καλλιεργούμε. Όλες αυτές οι πρακτικές αυξάνουν τις εκπομπές. Άδελφος κύριος Μαστάλκα για ένα λεπτό. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την εξαιρετική εργασία και συνεργασία. Συνεργαστήκαμε πολύ καλά για να φτάσουμε σε ένα συμβιβασμό κατά τον τριμερή διάλογο. Εδώ υπάρχουν και περιβαλλοντικά και κλιματικά στοιχεία γιατί όταν μιλάμε για την αποθήκευση ε, άνθρακα ε, πρόκειται για ένα τομέα ο οποίος έχει αμεληθεί και η χρήση της ε, υλοτομίας μέσα σε αυτή τη διεργασία θα οδηγήσει και σε δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Όμως δεν θα πρέπει να υπάρχει κακοδιαχείριση της δασοκομείας, γιατί θα περάσουμε από τις μονοκαλλιέργειες στη δημιουργία πολλαπλών ειδών. Κύριε Μαστάλκα, το λόγο έχει τώρα ο συνάδελφο Ρίχαρτ Ζέιμπερ από την Αυστρία για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και σα συγχαίρω για τα εξαιρετικά σα γερμανικά. Καλώ ορίζω ιδιαίτερω αυτή τη συμφωνία που ελπίζω να υπερψηφίσουμε αύριο. Νομίζω ότι επί της αρχής πρέπει να πούμε ότι σημαντικό στην πολιτική για το κλίμα είναι το βάρος να το φέρουν όλοι οι φορείς. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να συμπεριληφθεί και ο μέα του LULUCF. Γι' αυτό λοιπόν και θέτουμε κοινά πρότυπα σε ό,τι αφορά την υποβολή εκθέσεων για τα σχετικά πρότυπα. Επίσης, είναι σημαντικό να συνειδητοποιούμε ότι σε θέματα κλιματικής πολιτικής βρισκόμαστε στην αρχή μιας πορείας και γι' αυτό είναι βασικό οι αποφάσεις που έχουμε λάβει να εφαρμόζονται και να παρακολουθούμε πώς εφαρμόζονται. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο απλό αυτό όσο σε άλλους τομείς και γι' αυτό σημαντικό είναι να υπάρχουν κοινοί κανόνες όπως ορίζει στην δεύτερη έκθεση και να εξαγάγουμε τα απαραίτητα αποτελέσματα και θα πρέπει λοιπόν να αναλαμβάνουμε, να αναλαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα. Θα πρέπει να συνεχίζει να διαδραματίζει τον ηγετικό της ρόλο η Ευρωπαϊκή ε, Ένωση, αλλά είναι γεγονός ότι άλλα μέρη του κόσμου ευθύνονται και πολύ πιο πολλές εκπομπές. Ε, θα πρέπει να κοιτάξουμε λοιπόν ποιον πρώτο, ποιος θα είναι ο πρώτο στόχος μας προκειμένου να μπορέσουμε να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει για το μέλλον. Και επίσης ε, θα πρέπει να είμαστε ήρεμοι και σταθεροί και όχι να κάνουμε σπασμοντικές κινήσεις. Να δούμε ποιο είναι ο συγκεκριμένο αντίκτυπο των αποφάσεών μας. Και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να κοιτάξουμε αν είναι σωστέ οι αποφάσει μα, αλλά όπω είπα, να μην έχουμε σπανοδοτικέ κινήσει, να ακολουθήσουμε μία γραμμή ενιαία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τώρα το λόγο έχει η συνάδελφο Κρίστα Κλά, λέει ο πρόεδρο, Τα γερμανικά δύο λεπτά. Ευχαριστώ, πρόεδρε, επίτροπε, συνάδελφοι μπορούμε να, σε πολλά σημεία μπορούμε να διαφωνήσουμε για το ποιος είναι ο σωστός δρόμος για θέματα α, κλίματος. Αλλά εγώ πρέπει να πω ότι έχει καθυστερήσει κάπως ο ρυθμός μας ε, σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τομείς που δεν συγκαταλέγονται στο Λουλουσίεφ, σε ό,τι αφορά τα εθνικά κράτη, τα εθνικά ε, προγράμματα και τις σχετικές απαιτήσεις. Μέχρι το 2017 θα υπάρχει ένα νέο παγκόσμιο πρόγραμμα για το κλίμα και γι' αυτό δεν θα πρέπει να προαγάγουμε ένα σύστημα το οποίο δεν θα είναι ρεαλιστικό σε θέματα γεωργίας ιδιαιτέρως. Θα πρέπει σε παγκόσμιο επίπεδο να είμαστε αντικειμενικοί και θα πρέπει να προσέξουμε να μην δημιουργήσουμε ένα τέρας γραφειοκρατικό θέτοντας διαρκώς νέα πρότυπα τα οποία δεν θα μπορούμε να εγκαταλείψουμε στο μέλλον, στο περίπλοκο μοντέλο που έχουμε μπροστά μας για τον υπολογισμό των αερίων, άνθρα κτλ. Δεν υπολογίζεται ποιος θα είναι ο αντίκτυπος ε, Ποιο θα ήταν ο αντίκτυπο στην γεωργία, γιατί η γεωργία καλείται να επιτελέσει πολλέ λειτουργίε ε, έμεσα και άμεσα, τροφοδοτεί τον αυξανόμενο παγκόσμιο πληθυσμό και είναι ένα σημαντικό τομέας... κοινωνική αλλά και οικονομική ανάπτυξης. Αν επιβάλλουμε τέτοιες υποχρεώσεις για τον αγροτικό τομέα, πολλοί φαίνεται ότι ξεχνάνε ότι υπάρχουν και πολλά μικρά μέρη στον κόσμο που δεν είναι σε θέση να εκπληρώσουν όλους αυτούς τους όρους, τους περίπλοκους. Αυτό όμως ενδεχομένως να δημιουργήσει σε μία αντιστροφή των ε, καταστάσεων. Δεν ξέρω κατά πόσον όλα αυτά τα θέλουμε και τα χρειαζόμαστε. Εδώ βάζω ένα ερωτηματικό. Ευχαριστώ συνάδελφε Κλάς και τώρα καλώ τον ε, συνάδελφο Μπογκουσλάβ Σόνικ για ένα λεπτό να πάρει το λόγο. Ένα εναρμονισμένο σύστημα για την υποβολή αναφορών και τήρηση των επιδόσεων στις ε, εκπομπές του νανίου είναι κάτι το οποίο χρειάζεται. Θα πρέπει όμως βέβαια να είναι ε, καλά ρυθμισμένο το νομικό πλαίσιο. Όταν αποφασίσαμε να εγκριθεί ένα τέτοιο κανονισμό, είπαμε ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ε, από την πολυμορφία που κρατή στα κρατημέλη και τις διεθνείς επίσης υποχρεώσεις των κρατών για το Λούλου Σεφ. Θα πρέπει βέβαια να αποφύγουμε περιπλοκές, γραφειοκρατίες και επιπλέον διοικητικές δαπάνες. Θα πρέπει να δούμε πώς η ρύθμιση θα διέπεται από αναλογικότητα και λογική συνοχή. Θα πρέπει επίσης τα κρατημέλη να μην ενεργήσουν σε αντίθεση προς το διεθνές δίκαιο. Εγώ πάντως θεωρώ ότι είναι ε, λογικές οι τροπολογίες, ιδίως εκείνες που αποσκοπούν στο να δοθούν κάποιοι ορισμοί ε, σε σχέση με τα δάση. Διάει, το λόγο έχει συνάδελφος κυρία η, η συνάδελφος κυρία Τζόρντεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο μηχανισμός αυτός είναι κάτι το οποίο Σίγουρα χρειαζόμαστε. Θα πρέπει να υπάρξει εναρμόνιση, γιατί αν εναρμονιστεί το σύστημα αυτό, θα μειωθεί, αν θέλετε, το φορτίο που επιβαρύνει τις οικονομίες μας. Αλλά να προσέξουμε, γιατί θα πρέπει να μειωθεί και σε εθνικό επίπεδο το γραφειοκρατικό άχθος. Τα κρατημέλη ασφαλώς ε, κάνουν οικονομίες ε, σε ό,τι αφορά τέτοια θέματα διοικητικής ε, λειτουργίας. Να προσέξουμε, γιατί θα πρέπει να δαπανάμε πιο πολλά για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συμφωνώ με το κείμενο που αναφέρει ότι όλα τα μέσα αυτά θα πρέπει να είναι στοχευμένα. Όχι όμως μόνο το 50%. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερο ποσοστό. Δεν χρειάζεται να επενδύουμε μόνο σε αναπτυσσόμενες χώρες, γιατί αν προσπαθήσουμε να συλλέξουμε πιο πολλά χρήματα για το σκοπό αυτό, θα μπορούσαμε να να δημιουργήσουμε και πιο πολύ χάος σε τελική ανάλυση, γιατί τα κράτη-μέλη προφανώς θα ακολουθούσαν άλλα συμφέροντα και όχι μόνο θέματα κλίματος. Μικολάσικ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, Αυτοί οι μηχανισμοί θα συμβάλλουν στο να τηρούνται οι κανόνες για τη μείωση των εκπομπών. Έτσι θα τηρήσουμε, τόσο συμφωνήσαμε στο Κιώτο, έτσι θα πετύχει η Ευρωπαϊκή Ένωση τους στόχους της. Έτσι θα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος. Βεβαίως και οι καταθράσεις μεταφορές τώρα θα παρακολουθούνται. Γι' αυτό και σχετικές διατάξεις είναι πάρα πολύ καλοδεχούμενες. Όλα πρέπει να τα προσέξουμε στο μέλλον και θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια. Έτσι θα πρέπει να είναι δυνατόν να συγκρίνουμε τα δεδομένα από διαφορετικά κρατημέλη. Θα μπορούσαμε να έχουμε συγκεκριμένα μέτρα για τη μείωση των τελικά. Δίνω το λόγο στον συνάδελφο κύριο Γκρομπάλτσικ. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι πολιτικές για το κλίμα αποτελούν πολιτικές κλειδί για την ανάπτυξη της οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και βλέπουμε ότι στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός έναντι της από μετά από τις πολιτικές dumping στις χώρες αυτές και της έλλειψης κοινωνικής προστασίας μπορούν να περιορίσουν το κόστος παραγωγής με έναν τρόπο δυσανάλογο της Ευρωπαϊκής, με αυτόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ανταγωνιστική πλέον. Άρα, ο χώρος ανταγωνιστικότητας έχει να κάνει με το κόστος της ενέργειας. Κατανοούμε ότι οι καταστή. έχουν καταστεί ανταγωνιστικές ε, λόγω του συστολευτικού αερίου σε σχέση με τις χώρες της Απανατολής. Δεν θα πρέπει να θέτουμε παράλογες απαιτήσεις στις χώρες. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Διαφωνούμε με την προσέγγιση της αγοράς εργασίας στον τομέα ε, των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα που έχουν, ως επιπτώσει, που έχουν επιπτώσει θερμοκηπίου. Γι' αυτό δεν δεχόμαστε ότι μπορούμε να δεχτούμε αυτή τη λογική της αγοράς που θα μπορέσει να επιλύσει θέματα κλιματικών αλλαγών. Όμως μπορούμε να βελτιώσουμε τις γνώσεις μας ως προς τις χρήσεις της γης και του υπεδάφους. Η οργανική αυτή ύλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ροές ε, του άνθρακα, λαμβάνοντας υπόψη και καθαρά ανθρωπογενείς ε, παράγοντες. Πιστεύουμε ότι θα μπορούσαμε τουλάχιστον να πληρώσουμε τα χάσματα που έχουμε στον τομέα των γνώσεών μας. Ε, δίνω το, το λόγο στη συνάδελφο κυρία Έλενα Μπασέσκου. Ευχαριστώ. Η μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα έχει μεγάλη σημασία μέσω του μηχανισμού εποπτείας λοιπόν μπορούμε να κρίνουμε κατά πόσα απορροφούνται αυτά τα αέρια. Δέχομαι την πρόταση της Επιτροπής που βελτιώνει τις προδιαγραφές της Ένωσης που διέπουν το μηχανισμό. Επίσης, θα πρέπει να δούμε ποια είναι τα μέσα στον, που διαθέτουμε στον τομέα αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι μετά ε, έξι χρόνια της συμμετοχής της ε, Ρουμανίας στο ETS έχουμε τουλάχιστον 12.000 εγκαταστάσεις που έχουν μειώσει τις εκπομπές. Αυτό έχει μεγάλη σημασία για τη μείωση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα μέχρι ένα 20% μέχρι το 2020. Τελευταίος ομιλητής στη διαδικασία ΚΑΤΣΔΙΑ είναι ο συνάδελφος κύριος Έρικ Μπάνκι. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. Az üvegházhatású gázok kibocsátás csökkentése terén vállalt el. Η μείωση των εκπομπών αερίου θερμοκηπίου είναι κάτι το οποίο προαπαιτεί πολλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ποιο, πώς ε, ε, θα ορίσουμε το καθεστώς Λούλουσεφ, ιδιαίτερα όσον αφορά τη χρήση της γης. Θεωρούμε ότι οι δεσμεύσεις των κρατών μελών δεν επαρκούν. Γι' αυτό θα πρέπει να συμπεριλάβουμε άλλα, άλλες δυνατότητες, δηλαδή λογιστικά μέτρα και αλλαγές χρήσης η ανανέωση των δασών μπορεί να ε, έχει επιπτώσει σε συγκεκριμένα κράτη-μέλη όπως την Ουγγαρία. Θα πρέπει να ισχύσουν άλλα μέτρα λοιπόν για να λάβουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες ορισμένων κρατών μελών. Εξ της Επιτροπής δίνω το λόγο στην Επίτροπο, στην κυρία Χέντεγκαρντ. Θα είμαι σύντομη, Πρόεδρε γιατί ήταν τόσο θετικά όλα αυτά που άκουσα πώς επομένως υποστηρίζετε τις προτάσεις μας. Ε, ακούστηκε κάτι όσον αφορά την ανάγκη να βελτιώσουμε τη, γνώση μας. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω. Είναι απολύτως λογικό αυτό. Και τώρα έχουμε αρχίσει να, να ελέγχουμε. Αρχίσει να υπάρχει υποχρέωση λογοδοσία σε σχέση με το Λόλο Σεφ. Να αξιολογούμε τις επιπτώσει. Και γι' αυτό και είπαμε ότι έχουμε κάνει ένα το πρώτο βήμα. Είναι πολύ σημαντικό. Γιατί το επόμενο βήμα είναι ότι ο κόσμος θα θέλει να μάθει περισσότερα. Όλα αυτά αλληλοσυνδέονται. Να, επομένως πώς καταξιώνονται αυτό το νομοθέτημα που τώρα εγκρίνουν. Και μια φορά θεωρούμε ότι αυτές οι διεθνές ε, συναντήσεις μας κάνουν να αναρωτιόμαστε που καταλήγουν να καταλήγουν σε κάτι. Μα, να, ένα παράδειγμα πάρα πολύ χειροπιαστό. Θυμάστε πριν από 15 μήνες είχαμε βρεθεί στο Ντέρμπαν και κατόπιν είχαμε το κείμενο της Διεθνούς Συμφωνίας. Οπότε και τώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση όλα αυτά που προσπαθούμε να τα κάνουμε κοινοτικό δίκαιο. Όλα αυτά μπορεί να την διαφορά. Γιατί έχουμε τη Διεθνή Συμφωνία που άμα την κάνουμε εμείς νόμο θα ενεργοστούν και άλλοι να ακολουθήσουν. Να επομένω, ένα παράδειγμα του ότι πολλέ φορέ αυτέ οι βραδίε διαπραγματεύσει καταλήγουν σε κάτι το οποίο κάνει τη διαφορά στην ε, ζωή. Να επομένω, το πρώτο μου για τον Δούλεψα πολύ και ελπίζω ότι και αύριο θα ακουστεί πάρα πολύ θετική η φωνή του Κοινοβουλίου. Το λόγο έχει ο συνάδελφος κύριος Κρήτον Αρσένης για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Just some facts for colleagues to know. Κάποια στοιχεία για να πούμε στους συναδέλφους τι αποφεύγουμε για το αύριο. Η δραστηριότητα του Λούλου ε, ε, έχουν ως αποτέλεσμα οικονομία για τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Αν περάσουμε στο δεύτερο βήμα δε, μετρήσεις δηλαδή των εκπομπών Λουλουσιεφ σε ό,τι αφορά τους στόχους μας, θα έχουμε θετικό αντίκτυπο οικονομικό στα κρατη Άρα είναι προς το συμφέρον μας να κάνουμε όλοι τις ίδιες μετρήσεις και αυτό αποσκοπούμε με την νομοθεσία αυτή. Δεν υπάρχει οποιοδήποτε βάρος που να πέφτει πάνω στους αγρότες. Αυτό είναι σαφές το κείμενο και αποτελεί μικροστατιστικό εγχείρημα. Όπως είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά το 2020 θα έχουμε υποχρεωτικά λογιστικά πρότυπα σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες αυτές. Τι γίνεται μεταξύ του 2013 και μεταξύ 2020. Έχουμε μια προπαρασκευαστική φάση και υποχρεωτικές ε, τέτοιες ε, παροχές στοιχείων για κάθε χρόνο τα κράτη-μέλη μέχρι το 2020 θα πρέπει να ανακοινώνουν τις, ε, τους υπολογισμούς τους σε ό,τι αφορά τις ε, αγροτικές εκπομπές και στο τέλος της περίοδου αυτή θα πρέπει να ανακοινώσουν τις τελικές ε, τους τελικούς υπολογισμούς για κάθε έτος της περίοδου αυτής από το 2013 μέχρι το 2020. Μέχρι το 2020 λοιπόν θα ξέρουμε όλα τα λογιστικά είπα για όλη την περίοδο, περίοδο αυτή. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός σε σχέση με αυτά που είχαμε αποφασίσει όλοι στον Τέρμπαν και νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να είμαστε περήφανοι γιατί χάρη στις δύο αυτές εκθέσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδεικνύει σε όλο τον κόσμο πόσο δεσμευμένη είναι σε θέματα κλιματικής προστασίας. Έικουτ, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Νομίζω ότι έτσι μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση αυτή με σαφή λόγια ότι κάνουμε ένα μικρό βήμα όπως είπε και η Επίτροπος Χεντεγκάρτ. Ένα μικρό βήμα κάνουμε προς ε, την κατεύθυνση αυτή που αναφέρατε. Ένα μικρό βήμα. Διαπιστώνω κλείνοντας, ακούγοντας και τις παρατηρήσεις ε, εδώ στο, στην αίθουσα ότι όταν μιλάμε για κλίμα όλοι μας λένε ναι να πηγαίνουμε σιγά σιγά. Μου κάνει εντύπωση πόσο φοβόμαστε εδώ πέρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την κλιματική πολιτική. Μα σε λίγα πράγματα είναι τόσο ηγετική η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε μια ήπειρος που γυράσκει. Εξαρτόμαστε από εισαγωγές γιατί έχουμε λίγες πρωτεσίλες. Η οικονομία μας θα αναπτυχθεί λιγότερο γρήγορα από τη, της Κίνας, της Βραζιλίας και το εργασιακό κόστος είναι πολύ υψηλό και αυτή είναι η βασική εξήγηση για την υψηλή τιμή του ηλεκτρισμού. Και μετά τι θα πρέπει να καθόμαστε να περιμένουμε τι θα κάνει ο υπόλοιπος κόσμος. Θεωρώ ότι η μεγάλη μας ανταγωνιστικότητα προκύπτει από την καινοτομία μας. Καινοτομία σε μια καθαρή οικονομία. Και τώρα αν αυξήσουμε τις ε, κλιματικές μας φιλοδοξίες ε, μετά το 2020 θα δημιουργηθούν 6 εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας. Με τα βήματα αυτά λοιπόν κάνουμε ένα μικρό βήμα προς τα εμπρός, αλλά η καινοτομία η κοινοτομική ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα κυνηγάει το Κοινοβούλιο χωρίς να το φοβάται. Πολύ κύριε Έκουτ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ε, η συζήτηση κηρύσσεται περιοθήσα. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο στις 11.30 το πρωί. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη είναι οι παρεμβάσεις ενός λεπτού